της δημοκρατίας μας με μια ισχυρή ευρωπαϊκή δημοκρατία και το κοινοβούλιο αυτό θα είναι ένας βασικός φορέας αυτής της δημοκρατίας. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίε και κύριοι, έτσι ολοκληρώνεται η συζήτηση. Και επιτρέψτε μου παρακαλώ να προβώ μια συντομή ανακοίνωση που έχουν αναφέρει αρκετοί συνάδελφοι εντωμεταξύ. Έγινε μια επίθεση τρομοκρατική κατά της Αμερικανικής πρεσβείας της Βενγκάζης, όπου έχασαν τη ζωή τους και ο Αμερικανός πρεσβευτής και μέλη της οικογένειάς του αλλά και του προσωπικού της πρεσβείας και γι' αυτό θα ήθελα από τη θέση αυτή να απευθύνω τα θερμά συλληπιτήριά μας ε, στις αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών. Ευχαριστώ. έναρξη κυρίες και κύριοι συνάδελφοι έναρξη των ψηφοφοριών παρακαλώ διαδικαστικό ζήτημα παρακαλώ έχετε το λόγο Να υποστηρίξω αυτό το οποίο είπε ο Πρόεδρος μας για τα συλληπιτήριά μας στον Αμερικανικό λαό λόγω της επίθεσης στο προξενείο της Βενγκάζης όπου ε, σκοτώθηκε και ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρέπει επίσης να δώσουμε συλληπιτήρια και στο γενναίο λαό της Λιβύης που δεν του αξίζει η άσχημη αυτή εικόνα την οποία δημιουργούν ορισμένοι ακεραιόφρονες. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ανακοινώθηκαν στην Ολομέλεια αυτή τη Δευτέρα, τη 10η Σεπτεμβρίου, μία σύσταση της Επιτροπής Μεταφορών περί μη διατύπωση αντίρρησης σε εκτελεστικό μέτρο και μία σύσταση Επιτροπής Γεωργίας περί μη διατύπωση αντίρρησης σε κατεξιοδότηση πράξη. Δεν εκφράστηκε καμία αντίρρηση στις στάσεις αυτές εντός της 24 ώρης προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 87α του κανονισμού. Συνεπώς, οι συστάσεις αυτές θεωρούνται εγκριθήσεις με ισχύ από την 11η Σεπτεμβρίου 2012 και οι αποφάσεις θα δημοσιευθούν σε κείμενα που εγκρίθηκαν τη σημερινή συνόδου. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Κύριε Έλερ, έχετε το λόγο. Um, um, Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και ως πρόεδρος της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και εξ όλων των εδώ παρόντων, παρόντων να απευθύνω